κυρίε και κύριοι, να σα καλωσορίσω στη σημερινή συνεδρίαση τη αντιπροσωπεία μα για τη σχέση με την Κεντρική Αμερική. Να καλωσορίσω τον πρέσβη τη Γουατεμάλα, τον κύριο Γουτιέρε, τον πρέσβη του Πελίζε, κύριο Βέρνον, τον πρέσβη τη Κωνσταντίνα, κύριο Αλφάρο. επίση περιμένουμε τον κύριο Πόνζ από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, προϊστάμενη τη Υπηρεσία Εξωτερική δράση, ο οποίο θα έρθει σε λίγο. Η διερμηνία παρέχεται στις, στα αγγλικά, ισπανικά, ελληνικά και στα γαλλικά. Το σχέδιο της μερίσιας διάταξης έχει διανεμηθεί στα αγγλικά, ελληνικά και στα ισπανικά και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα θεωρηθεί ότι η μερίσια διάταξη εγκριθεί. Όπως γνωρίζετε, στις 19 Απριλίου του 2018 ο κύριος Κανέλ ορκίστηκε επισήμως σαν νέος πρόεδρος της Κούβας έπειτα από μια μυστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Συνέλευση της χώρας ο διάδοχος του κυρίου Κάστρο έλαβε στην ψηφοφορία 603 από τις 604 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 99,38% της Αθνοσυνέλευσης... εξασφαλίζοντας πενταετή προεδρική θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι έχω αποστείλει συγχαρητήρια επιστολή στον κύριο Κανέλ, την οποία μπορείτε να βρείτε στο φάκελο που σα έχει διανεμηθεί. Παραπέρα και σε σχέση με την Ικαράγουα, θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου για τι πρόσφατε εξελίξει στη χώρα, όπου οι διαμαρτυρίες κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος είχε σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον 30 θανάτους. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που τέθηκαν σε ισχύ την 16η Απριλίου έχουν σαν στόχο μεταξύ άλλων την διάσωση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων προβλέποντας τη μείωση των συντάξεων κατά 5% και αύξηση των εισφορών των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους. Στις 22 Απριλίου ο πρόεδρος Ορτέγκα παραδέχθηκε ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι βιώσιμες, ανακοίνωσε την κατάργησή τους και κάλεσε όλες τις πλευρές για έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο. Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο σεβασμιότατος καρδινάλιος Μπρένες και οι επίσκοποι της επισκοπικής διάσκεψης στην Καράγουα αποδέχθηκαν να συμμετάσχουν ως μεσολαβητές και μάρτυρες στον διάλογο που κάλεσε ο πρόεδρος Ορτέγκα. Απευθύνουμε έκκληση για τον τερματισμό της βίας, και προτρέπουμε όλα τα μέρη να λάβουν μέρος στο διάλογο αυτό και σημαίνει στον φάκελό σα, θα βρείτε μια δήλωση της, Επιτροπή, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης εκ μέρους της κυρίας Φαντερίκα Μονκερίνη σχετικά με τα γεγονότα που συνέβησαν στην Ικαράγουα. Η αντιπροσωπεία μας σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στη χώρα. Στο σημείο 3 που αφορά στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα αποτελέσματα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το σημείο 2 και το γεγονός ε, του θέματος της Νικαράγουα, ε, νομίζω ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να καταδικάσει την ε, καταπίαση που βίωσε η Νικαράγουα τις τελευταίες ημέρες, όπως πολύ σωστά είπε η Πρόεδρος, πάνω από 30 νεκρούς. Και εγώ πραγματικά πιστεύω ειλικρινά ότι η πρόεδρος εξ ονόματος αντιπροσωπείας μας, ε, όπως και όταν ε, ε, πέθανε ο Φιντέλη Κάστρο, έστειλε σωστά συγχαρητήρια επιστολή στο νέο ε, πρόεδρο τώρα θα πρέπει να στείλει μια επιστολή για να καταδικάσει τα γεγονότα και να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς ε, τα οικογένειε των θυμάτων. Οι χώρες ε, της περιοχής ήδη εξέφρασαν την άποψή της στην ομάδα Λίμα και θέλω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως κάνουμε πάντα που καταδικάζουμε οποιαδήποτε πράξη καταπίεσης, να κάνουμε το αντίστοιχο και για τα όσα συνέβησαν στην Ικαράγω. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη η παρατήρηση. Πάμε στο σημείο 3, όπου αφορά στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματο που πραγματοποιήθηκε στην Γουατεμάλα την Κυριακή στι 15 Απριλίου του 2018, αναφορικά με την επίλυση τη συνοριακή σύγκρουση με τον Μπελίζ. Στι 15 Απριλίου, λοιπόν, διεξήχθη δημοψήφισμα με αντικείμενο την επίλυση τη εδαφική διαμάχη ανάμεσα στον Μπελίζ και στην Γουατεμάλα. Οι ψηφοφόροι ρωτήθηκαν για το αν η κυβέρνηση της Γουατεμάλα θα πρέπει να ζητήσει από το Διεθνές Δικαστήριο να επιλύσει επιτέλους την εδαφική διαμάχη ως προς την δέσμευση που υπεγράφει τον Δεκέμβριο του 2008 μεταξύ της Γουατεμάλα και του Μπελίζ. Η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων με ποσοστό 95,88% ψήφισε υπέρ της παραπάνω πρότασης. Εν συνεχεία, το Μπελίζ θα πραγματοποιήσει με τη σειρά του παρόμοιο δημοψήφισμα για το εν ζήτημα, αν και ακόμη δεν έχει καθοριστεί επίσημα κάποια ημερομηνία. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να δώσω τον λόγο στην αυτοεξοχότητα πρέσβη τη Γουατεμάλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριο Γκουτιέρε, για να μας πει τη δική του τοποθέτηση. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να μοιραστώ μαζί σας με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις ε, με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος που έγινε στις 15 Απριλίου στη Γουατεμάλα. Εδώ και πάνω από 150 χρόνια υπάρχει μια διαφορά ε, μεταξύ της δημοκρατίας της Γουατεμάλας που θεώρησε ότι είναι θέμα του κράτους, καταρχάς με το Ηνωμένο Βασίλειο και την ε, Μεγάλη Βρετανία και τη Βόρεια Ιρλανδία και με την έναρξη των διπλωματικών σχέσεων στις 11 Σεπτεμβρίου του 1991 πλέον με τον Πελής. Και εκεί ε, Υπάρχει το θέμα της ε, αναγνώρισης εδαφών που βρίσκονται υπό διοίκηση της, ε, του Μπελής. Καθώς επίσης ε, και να εξαντλήσει και όλα τα μέσα που είχε στη διάθεσή της για την επίλυση των διαφορών, όπως για παράδειγμα επιστολή προς τα Ηνωμένα Έθνη και μέσω του Διεθνούς Δικαίου, η Γατεμάλα και το Μπελής αποφάσισαν με σύσταση του Γενικού Γραμματέα της Οργάνωσης των Αμερικανικών Χωρών να προσφύγουν στο δικαστήριο, στο Διεθνές ε, δικαστήριο για να λύσουν οριστικά τη διαφορά μεταξύ τους. Αυτή η δέσμευση περιλαμβάνεται στην ε, ειδική συμφωνία μεταξύ Γουατεμάλας και Μπελής ε, για την επίλυση του εδαφικού, νησιωτικού και θαλάσσιου θέματος της διαφοράς μεταξύ Γουατεμάλας και Μπελίσε στο Διεθνές Δικαστήριο. Αυτό έγινε στις 8 Δεκεμβρίου του 2008. Μετά, μετά από ένα πρωτόκολλο που υπεγράφει στις 25 Μαΐου του 2015 στην Γουατεμάλα, οι δύο χώρες αποφάσισαν να ξεκινήσουν ε, δημοψηφίσματα είτε ταυτόχρονα είτε ξεχωριστά ε, σε ημερομηνίες που αρμόζουν στην κάθε πλευρά. Αυτή η ειδική συμφωνία και το σχετικό πρωτόκολλο επιτρέπουν επίσης ε, να τηρηθεί αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 19 των μεταβατικών και τελικών διατάξεων της ε, του συντάγματος της ε, Δημοκρατίας της Βατεμόλα, που καθορίζει ότι η κυβέρνηση της Γουατεμάλας έχει αρμοδιότητα για να επιλύσει τα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα της Γουατεμάλας έναντι του Μπελής ε, που αφοράουν και τα εθνικά συμφέροντα και οποιαδήποτε οριστική συμφωνία θα πρέπει να περάσει και από μια διαδικασία δημοψηφίσματος. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσω ότι αυτός ο συνταγματικός ε, κανόνας προβλέπει ότι η κυβέρνηση της Γουατεμάλας θα προωθήσει κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις με, την, ε, με τον Πελής ε, και όσον αφορά τα θέματα της υποκότητας οι ε, κάτοικοι του Μπελίσια θα χαίρουν του ίδιου καθεστώτος που ισχύει και για όσους ε, προέρχονται από χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Γι' αυτό ακριβώς και από το 2005 η Γουατεμάλα ε, προσπαθεί να υπάρχει μια ξεχωριστή επίλυση μεταξύ των διμερών σχέσεων και της διαφοράς που υπάρχει στα εδαφικά και προσπαθεί να δημιουργήσει μια φυσική και δυναμική σχέση η οποία θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην ευγένεια και στη συνεργασία με τον Μπελίσια. Αυτή η θετική στάση μας επέτρεψε να εργαστούμε επικοδομητικά στις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε, κυρίως μετά από τα περιστατικά τα οποία υπήρξαν στην περιοχή της Αδιασένσα, την Πράσινη Γραμμή, καθώς επίσης και την υπογραφή ε, των συμφωνών της Πλαθένθειας στις 14 Δεκεμβρίου του 2014, που έχουν ως στόχο να ενδυναμώσουν τη διμερή σχέση, ιδίως ε, σε θέματα που ενδιαφέρουν και προσεγγίζουν περισσότερο τους δύο λαούς ε, μπορούμε να πούμε ότι η σχέση μας με τον Μπελής ε, ορίμασε σε μεγάλο βαθμό και οι δύο λαοί και οι κυβερνήσεις. Ε, δεν ζούμε με την πλάτη γυρισμένα τον άλλον, αλλά προωθούμε με θετικό τρόπο και επικοδομητικό τρόπο μεγαλύτερα επίπεδα προσέγγισης. Σε συνέχεια το προηγουμένο, στις 23 Οκτωβρίου του 2017, το ανώτατο εκλογικό ε, δικαστήριο κάλεσε τους πολίτες της Γουατεμάλας ε, σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες ε, να ψηφίσουν σε ένα δημοψήφισμα για να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά στην εξή ερώτηση την οποία διατύπωσε το Κογκρέσο της Δημοκρατίας όπως προβλέπει και η Ειδική Συμφωνία. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε νομική απέτηση της Γουατεμάλας κατά του Μπελής όσον αφορά ε, υπηρετικά και νησιωτικά εδάφη και τις αντίστοιχες ε, θαλάσσιες περιοχές και χωρικά ύδατα θα υποβάλλονται στο ε, Διεθνές Δικαστήριο προκειμένου να επιλύσει οριστικά και ότι αυτό θα καθορίσει τα σύνορα των περιοχών των δύο πλευρών. Μετά από αυτή την πρόσκληση ε, υπήρξε και μια εκστρατεία ενημέρωση ε, στο υψηλότερο επίπεδο. Επικεφαλήθηκαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος ε, ηγήθηκε των προσπαθειών για να ενημερώσουμε τους πολίτες για την ιστορική ευκαιρία να ληφθεί μια απόφαση η οποία θα μας οδηγήσει σε μια οριστική λύση για τι κοινέ προκλήσει που έχουμε με τον Πελή. Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση της Γουατεμάλα σε ενημέρωσε τις διάφορες πλευρές και τους διάφορα τμήματα της κοινωνίας της Γουατεμάλας για το θέμα και τις πιθανές λύσεις για την επίλυση της διαφοράς μας. Στις 15 Απριλίου του 2018, που ήταν η ημερομηνία που καθορίστηκε για το δημοψήφισμα, χάρη στα μέτρα ασφαλείας ε, τάξεως, καθώς επίσης και τις δράσεις που έγιναν σε όλα τα κέντρα ε, τα εκλογικά, ε, το δημοψήφισμα διεξήχθη ειρηνικά και χωρίς προβλήματα. Θα πρέπει επίσης να πούμε πώς οι τρεις αρχές του κράτους ε, ε, δήμοι, ε, περιφέρειες, κοινωνικοί και επιχειρηματικοί ιδέτες, καθώς επίσης και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και τη βοήθειά τους προκειμένου να οργανώσουμε και να ζήσουμε μια ιστορική ημέρα στην πολιτική ζωή της Βατεμάλας. Μια ημέρα με την οποία ε, βάσει των προκαταρκτικών στοιχείων ε, του εκλογικού δικαστηρίου ασκώντας ε, την κυριαρχία του, ο λαός της Βατεμάλας αποφάσισε να τεθεί το θέμα της εδαφικής, νησιωτικής και θαλάσσιας διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο με μια πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία της τάξης του 95,88%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι επειδή δεν ήταν υποχρεωτική η ψήφο, η συμμετοχή ε, άνω των 2 εκατομμυρίων ατόμων, δηλαδή 26,65% σε αυτό το δημοψήφισμα, ξεπέρασε όλες τις προσδοκίε. Πιο συγκεκριμένα, αν λάβουμε υπόψη τα αποτελέσματα των δύο δημοψηφισμάτων που έγιναν στο παρελθόν, που είχαν ε, πολύ μικρότερο ποσοστό συμμετοχής 15% στο δημοψήφισμα για συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του 1994 και 18,55% στο δημοψήφισμα για τις ε, ειρηνευτικές συμφωνίες του 1999. Άρα, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ε, της 15ης Απριλίου αποτελεί ιστορικό και νόμιμο αποτέλεσμα της δημοκρατικής έκφρασης του λαού της Γουατεμάλας και επιβεβαιώνει και πάλι τη δέσμευσή μας ότι θέλουμε να αναζητήσουμε μια ειρηνική και οριστική λύση στη διαφορά που υπάρχει σε εδαφικά, νησιωτικά και θαλάσσια ζητήματα με τον Πελής και όσον αφορά τα όσα έχει δεσμευτεί να κάνει η Γουατεμάλα σε διεθνέ επίπεδο. Εδώ δεν θα πρέπει να ξεχάσω να αναγνωρίσω και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωση μέσω του προγράμματος ε, προώθησης και συμμετοχής των πολιτών στο δημοψήφισμα με ένα ποσό της τάξης των 114 εκατομμυρίων ευρώ και να ευχαριστήσω επίσης ε, και την ε, δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16 Απριλίου, καθώς επίσης και τη δέσμευσή της να υποστηρίξει πρωτοβουλίες για την εξέλιξη της περιοχής της Αδιασένσια, που να ευχαριστήσω επίσης και την βοήθεια που λάβαμε από την ομάδα φίλων. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι όταν θα έχουν ολοκληρωθεί και τα τυπικά για την επισημοποίηση των αποστελεσμάτων ε, του εκλογικού δικαστηρίου, το δικαστήριο θα πρέπει να ανακηρύξει επισήμω τα αποτελέσματα και να κοινοποιήσει το Κογκρέσο της Δημοκρατίας, ώστε να τα διαβιβάσει και αυτό με τη σειρά του στην κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή ολοκληρωθεί λοιπόν αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει να κοινοποιήσουμε στο Διεθνές Δικαστήριο και στην κυβέρνηση του Μπελίζ την δημοκρατική και κυρίαρχη απόφαση του λαού της Βατεμάλας ε, για να ξεκινήσει η διαδικασία για την οριστική λύση αυτής της ε, διαφοράς. Ολοκληρώνω επαναλαμβάνοντα ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Γουατεμάλας και Μπελίσα περνούν ε, αυτή τη στιγμή την καλύτερη στιγμή τους και η κυβέρνηση τη Γουατεμάλας θα προσπαθήσει να ενισχύσει τους δεσμούς φιλίας που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός του Μπελίζ, ο κ. Διν Μπαρό, τον πρόεδρο τη Γουατεμάλας, ε, δεν θα πρέπει να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας τα προβλήματα που κληροδότησαν οι πατέρες μας εμάς. Η Γουατεμάλα λοιπόν ε, με αυτό το ίδιο πνεύμα ε, θα αντιμετωπίσει την αδερφή χώρα και την κυβέρνηση του Μπελής και θα προχωρήσει και αυτή με τη σειρά της στο δημοψήφισμα βάσει του άρθρου 7 της Ειδικής Συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρέσβη και τώρα να δώσω τον λόγο στην αυτοεξοχότητα πρέσβη τον κύριο Thank you, uh, Madam Chair, for the... Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απίθυνε η αντιπροσωπεία σας. Να σας μιλήσω σήμερα για τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στη Γουατεμάλα που έλαβε χώρα στις 15 Απριλίου του 2018. Επίσης να ευχαριστήσω τον συνάδελφο πρέσβη της Γουατεμάλας για, τα, για την πολύ καλή ενημέρωση. Η κυβέρνησή μου ήταν από τις ε, πρώτες που συνεχάρει την κυβέρνηση και το λαό της Δημοκρατίας της Γουατεμάλας για το ειρηνικό και επιτυχημένο δημοψήφισμα που βασίζεται στην Συμφωνία των Δύο Χωρών του 2008 το δημοψήφισμα της Γουατεμάλας από τη δική μας οπτική γωνία αποτελεί ιστορικό γεγονός. Και το συντριπτικό ναι είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα στον δρόμο προς την ειρηνική επίλυση ε, των ε, απαιτήσεων της ε, Γουατεμάλας. Τα νέα είναι πάρα πολύ θετικά, λοιπόν. Από τη δική μας πλευρά, εκ μέρους της κυβέρνησής μας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι το, το Μπελίζε έχει δεσμευθεί να διεξάγει το δικό του ε, δημοψήφισμα σύμφωνα με ε, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Wilfred P. Έρνικτον σας ενημέρωσε τον Δεκέμβριο του 2017 ότι το Μπελίζε θα διεξάγει το δημοψήφισμά του μετά από την ε, απαιτούμενη εκ του συντάγματος επανακαταγραφή των ψηφοφόρων. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους και μόλις ολοκληρωθεί το Μπελίζε θα διεξάγει το δημοψήφισμά του. Ταυτόχρονα το Μπελίζ ε, εντατικοποιεί ακόμα περισσότερο πλέον την δική του ε, εκστρατεία ενημέρωσης της ε, κοινωνίας έτσι ώστε όλοι οι ψηφοφόροι να είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι όταν κληθούν να απαντήσουν στο ίδιο ερώτημα που απάντησαν και οι πολίτες της Ουατεμάλας περί παραπομπής της διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την συνεχιζόμενη υποστήριξή της στη διαδικασία ε, συμπεριλαμβανομένης και της ε, χρηματοδότησης που παρέχει. Το Μπελίζ επαναλαμβάνει την ανάγκη ε, το γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραμείνει στην ενδιάμεση ζώνη και να συνεχίσει να χρηματοδοτεί με επαρκής πόρους τη διαδικασία ε, ανεξάρτητα και αμερόληπτα. Ε, προσβλέπουμε σε συνεχιζόμενη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη και τα, τα κράτη της ε, ομάδας των φίλων. Η, όσο η διαδικασία συνεχίζεται, το Μπελίζε εξακολουθεί να κάνει προσπάθειες να εμβαθύνει και να βελτιώσει τις σχέσεις του με τη γειτονική Γουατεμάλα ιδιαίτερος ε, κατόπιν μιας πρόσφατης υπουργική συνάντησης μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών η, δημιουργήθηκε, μάλλον επαναδραστηριοποιήθηκε η Επιτροπή Μπελίζε Γουατεμάλα τον περασμένο μήνα. Αυτή η κοινή επιτροπή θα ξανασυνέλθει σύντομα για να προωθήσει την συνεργασία και τις σχέσεις καλής γειτονίας και να συνεχίσει να ε, εργάζεται στην εφαρμογή των 14 σημείων που έχουν συμφωνηθεί, 14 τομέων συνεργασία. Ω μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, η, το Μπελίζε θέλει να συνεργαστεί με τη Γουατεμάλα για την ανάπτυξη ενό μηχανισμού ε, τέτοιων μέτρων ε, οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Ε, ε ιδιαίτερα στην περιοχή των νότιων συνόρων του Μπελίζα με τη Γουατεμάλα για να αποφύγουμε τις εντάσεις και ενδεχόμενα επεισόδια Θέλουμε ότι αυτά, ε, πιστεύουμε ότι αυτά τα μέτρα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Συνεπώς, ε, εν ώψη ε, ε μιας του θέματος από το Διεθνές ε, Δικαστήριο, το Μπελίζε είναι προσιλωμένο στις φιλικές σχέσεις με τη Γουατεμάλα, τίνουμε χειραφιλίας και επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας ε, να διεξάγουμε το δικό μας δημοψήφισμα το συντομότερο δυνατό. Μία ακόμα φορά θα ήθελα να συγχαρώ την κυβέρνηση και το λαό της ε, Γουατεμάλας για την επιτυχή διεξαγωγή του δικού τους δημοψηφίσματος. Βρισκόμαστε ένα ακόμα βήμα πιο κοντά σε μία ακόμα ιστορική μάλλον ευκαιρία να επιλύσουμε ειρηνικά μία, ένα από τις, μία από τις τελευταίες ε, διαφορές που υπάρχουν στην Κεντρική Αμερική. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Να καλωσορίσω τον κύριο Πόνς και να του δώσω αμέσω το λόγο για να μας ενημερώσει και εκείνος που Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε για να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας ενδιαφέρει πολύ και είμαι πολύ ικανοποιημένο που μπορώ να συγχαρώ καταρχάς ε, τη Γουατεμάλα, το φίλο μας τον πρέσβη της Γουατεμάλας ε, και όλη τη Γουατεμάλα για τη διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος που αποτελεί ένα βήμα το οποίο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ιστορικό για την επίλυση μιας διαφοράς πάρα πολύ δύσκολης ε, με ειρηνικά μέσα τα οποία συμφώνησαν και οι δύο πλευρές και τα οποία βασίζονται στο διάλογο είναι ουσιαστικά το DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω, να επιλύει τέτοιες διαφορές με τέτοιο τρόπο ή τουλάχιστον να κάνει ό,τι μπορεί και για άλλη μια φορά να συγχαρώ τη Γουατεμάλα ε, για αυτή την προσπάθεια που έκανε και γνωρίζουμε πόσο δύσκολο υπήρξε. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ και τον Μπελίζε και τον ε, φίλο μας τον πρέσβη του Μπελίζε για την επαναλαμβανόμενη δέσμευσή του να διεξάγουν και αυτοί το δημοψήφισμα το συντομότερο δυνατόν. Ε, νομίζω ότι αυτό μας είπε και πραγματικά ε, εμπιστευόμαστε τα όσα μας λένε και πιστεύουμε ότι θα γίνει όσο το συντομότερο γίνεται γιατί έχει ξεκινήσει μια διαδικασία και πιστεύω ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την όθηση που έχει δοθεί ε, μέσω αυτού του δημοψηφίσματος. Εμείς και εγώ προσωπικά είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ την περιοχή της Αντιασένσια, της πράσινης γραμμής μεταξύ των δύο χωρών και να δω πραγματικά τις προσπάθειες που κάνουν και οι δύο πλευρές και την επανέναρξη της Μικτής Επιτροπής Γουατεμάλας Μπελίσε, την επιστροφή των πρέσβεων, όλα αυτά είναι ε, θετικά στοιχεία και ε, θα ήθελα επίσης να πω και κάτι το οποίο δεν λέγεται πολύ συχνά αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. αυτή η όθηση, αυτή η δυναμική μπορεί να αποτελέσει και παράδειγμα για άλλες ε, διαφορές και συγκρούσεις. Η κάθε μία βέβαια είναι διαφορετική, δεν προσπαθούμε να κάνουμε καμιά μορφής προσωμείωση, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά και θεωρώ ότι ο αντίκτυπο είναι θετικό πέραν τη Γουατεμάλα και του Μπελίζε. Εάν λοιπόν στο τέλο της πορεία υπάρξει μια συμφωνία όπω ελπίζουμε και να αποφασθεί το διεθνέ Δικαστήριο ε, γιατί και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει, πιστεύω ότι θα δημιουργήσουν ένα πολύ καλό προηγούμενο. Η συμφωνία των δύο πλευρών είναι πάρα πολύ ικανοποιητική και βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ καλό συντονισμό μεταξύ Γουατεμάλα και Μπελίζια και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να επιληθεί οποιαδήποτε διαφορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε από πολιτική σκοπιά πολύ στεναρά την όλη πορεία αλλά και με χρηματοοικονομική βοήθεια, με τη στήριξη που προσφέραμε στο γραφείο της Οργάνωσης των Αμερικανικών Χωρών και στην περιοχή της Διασένσια εδώ και πάρα πολύ καιρό και ε, ελπίζουμε να συνεχίσει η συνεργασία και να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τη συνέχιση αυτής της διαδικασίας μέχρι να φτάσουμε σε μια ειρηνική λύση. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίω ότι πρόκειται για μια προσπάθεια η οποία ε, σε ιδανικέ συνθήκε θα πρέπει να υποστηριχθεί και από άλλε πλευρέ, αλλά ίσω αυτό να είναι το επόμενο κεφάλαιο. Αυτό το οποίο θέλουμε να επισημάνουμε σήμερα είναι τη συμφωνία και την ε, υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στο παρελθόν και τώρα αλλά και στο μέλλον. Για άλλη μια φορά λοιπόν σα ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία. Και εγώ σας ευχαριστώ και να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο στην Κρίματα. Muchas gracias, Presidenta. Evidentemente, muchísimas gracias a los dos embajadores por las Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εξηγήσεις του τους δύο πρέσβεις και την υπηρεσία εξωτερικής δράσης της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαίρομαι πάρα πολύ που γίνονται βήματα, που βλέπω έναν ειλικρινή, μια ειλικρινή πρόθεση διαλόγου για τους καινούριου διάβλους επικοινωνίας και για τις ε, προσπάθειες που καταβάλλονται να φτάσουμε σε μια οριστική συμφωνία αυτού του, αυτής της ιστορικής ε, διαμάχης. Ο, έχετε όλοι μας την υποστήριξη και οτιδήποτε χρειάζεστε από την πλευρά μας. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Γουατεμάλα είναι εντυπωσιακό Η συμμετοχή με τα δικά μας πρότυπα είναι βέβαια πολύ χαμηλή, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ψηλότερη από τη συμμετοχή σε προηγούμενα δημοψηφίσματα. Συνεπώς θα πρέπει να μας χαροποιήσει ακόμα και η συμμετοχή, το ποσοστό. Και πολύ δε περισσότερο που και το Μπελίζ έχει σκοπό να διεξάγει το δικό του δημοψήφισμα. Όλα αυτά πολύ καλά. Αλλά θα πρέπει... Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να είναι ανησυχητικό. Και αυτό είναι η επόμενη μέρα το αποτέλεσμα, το του δημοσιογράφου στον Πελίζη μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό. Αν είναι θετικό, όλα καλά. Ανοίγει ένας καινούριο ε, δρόμος. Ας πούμε ότι, ότι, ότι εντάξει, η τελική ενα καινουριο δρομος α πουμε οτι οτι μπορεί να μην βρεθεί τόσο εύκολα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι μια καλή εξέλιξη το ναι στον Πελίζε. Αν όμω στον Πελίζε το δημοψήφισμα δώσει όχι, τότε τα πράγματα θα περιπλακούν. Ποια θα ήταν τα επόμενα βήματα τα οποία θα κάνατε. Αν η κυβέρνηση του Μπελίζε ε, κάνει ε, εκστρατεία υπέρ του ναι, τι θα γίνει αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Προφανώ το δημοψήφισμα διοργανώνεται δημοκρατικά, αλλά ποια θα είναι η θέση της κυβέρνηση μετά. Είναι προφανέ ότι ε, θα έχει άμεση επίδραση ε, πάνω στην ίδια την κυβέρνηση το ένα ενδεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα. Αυτά. Και, και πάντως έχετε την πλήρη μας στήριξη. κύριε Πρέσβη, θα ήθελα να σα ρωτήσω αν θέλετε να απαντήσετε στην ερώτηση που ο κύριο Μάτο σα έθεσε. Thank you for, for the question. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις και κυρίως ε, για την ε, συνεχή στήριξή σας. Θα πρέπει να είναι σαφές ε, διότι, ότι η πάγια θέση της κυβέρνησης του Μπελίζε είναι ναι ε, στην προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο. Και η θέση της κυβέρνησης ήταν ε, η ίδια ε, και σε, από διάφορα πολιτικά κόμματα εδώ και αρκετό καιρό. Επομένως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε επίπεδο κυβέρνησης επιθυμούμε μια καταφατική ψήφο για να μπορέσουμε να προσφύγουμε στο δικαστήριο. Όσον αφορά τα πλαίσια μιας ε, ε, δημοκρατίας η οποία λειτουργεί με δυναμικό τρόπο θα είναι μια δυναμική εκστρατεία για να μπορέσουν να αποφασίσουν αυτοί οι οποίοι επιθυμούν να πούν ναι και αυτοί που επιθυμούν να πούν όχι. Η παρούσα θέση της κυβέρνησης όσον αφορά την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού είναι να δώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες ε, στο κοινό του Μπελίζη όσον αφορά το ιστορικό του, του θέματος και τους διάφορους ισχυρισμού ε, και το αίτημα και φυσικά να ε, επιταχύνουμε και την ημερομηνία του δημοψηφίσματος. Το θέμα αυτό αυτή τη στιγμή είναι το πιο σημαντικό πολιτικό και διεθνές ζήτημα για τον Μπελίζε. Θα γίνει μια μακρά συζήτηση και αναμένουμε ότι αυτή τη στιγμή γίνει το δημοψήφισμα, θα υπάρχει ε, μεγάλο ποσοστό συμμετοχής. Αυτά μπορώ να απαντήσω προς το παρόν στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ και κάτι τελευταίο βέβαια. Δεν έχουμε καν διανοηθεί σε επίπεδο κυβέρνηση ε, τι θα συμβεί σε περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική, γιατί είναι τόσο ε, βέβαια η κυβέρνηση ότι το επόμενο βήμα είναι η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και να σας ευχαριστήσω και εγώ από τη θέση της Πρόεδρου και για την ενημέρωση αλλά και για τις, εξελι... εξηγήσεις που δώσατε. Να σας διαβεβαιώσω ότι η αντιπροσωπεία μας θα παρακολουθεί τις προσπάθειες στενά για το, ε, επερχόμενο δημοψήφισμα και βεβαίως προσωπικά εύχομαι να δοθεί οριστική λύση, ειρηνική όπως είπατε, και που όπως επίσης είπατε θα ενισχύσει τους δεσμούς φιλίας των ε, δύο λαών. Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, στο τέταρτο, που αφορά στα συμπεράσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Παρλασέν και του Παρλασέν που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου του 2018 στην πόλη του Παναμά στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της μόνιμης επιτροπής Eurolat. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της συνεδρίας της Eurolat στην πόλη του Παναμά στις 5 Απριλίου του 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας του Παρλασέν με επικεφαλή στον κύριο Φαρινόνη και αντιπροσωπείας στην ΔΕΚΑΜ με επικεφαλή στον αντιπρόεδρο της ΔΕΚΑΜ, τον κύριο Γκαβριέλ Μάτο. Το κύριο θέμα της συζήτησης αφορούσε στους κανόνες διαδικασίας της μελλοντική Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, τους οποίους, όπως γνωρίζετε, συζητάμε με τους εταίρους μας εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια. Από την ενημέρωση που είχα, η συνάντηση ήταν πολύ αποτελεσματική, όπου έγινε προσπάθεια να βρεθεί διέξοδος για την σύσταση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεντρικής Αμερικής. Υπήρξαν καλές συζητήσεις για την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Αμερικής και για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Αμερικής. Και δεν υπάρχει καμία αναφορά αρνητική. Αλλά θα ήταν να δώσω καλύτερα το λόγο στον Αντιπρόεδρο που εκπροσώπησε και την Επιτροπή της ΔΕΚΑ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι έγινε αυτή η συνεδρίαση την τελευταία ημέρα της συνόδου της Eurolat και το πρώτο το οποίο θα ήθελα να κάνω είναι να ευχαριστήσω δημοσίως ε, τους αμφιτριονές μας ε, οι οποίοι όπως πάντα μας έκαναν να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Τα βασικά σημεία της συζήτησης, ε, τα πρώτα τα είπε η Πρόεδρος, ε, ο κανονισμός της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΣΥΚΑ και επίσης η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντρικής Ενεργικής. Όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΣΥΚΑ, Έγινε μια εξαιρετική παρουσίαση του υπευθύνου διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο, του Τζοβάνι Ντιτζιρόλαμο, και επίσης ε, μας είπε κάποια πράγματα για το υποπεριφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Αμερική, που είχε μεγάλη σημασία εδώ και κάποιο καιρό, και για το 2020 θα έχει μια αύξηση και θα φτάσει μέχρι και τα 120 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό, το οποίο ήταν 95 εκατομμύρια, επομένω έχουμε μια αύξηση της τάξης του 30%. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, ε, και αυτό είναι πολύ χρήσιμο και εμεί θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παραμείνει, σε τέσσερα σημεία. Οικονομική ολοκλήρωση, κράτος δικαίου και ασφάλεια, κλιματική αλλαγή και κυρίως διαχείριση των καταστροφών και ε, επισητιστική ασφάλεια. Ε, υπάρχουν ε, περίπου 11 προγράμματα τα οποία είναι υπό εκτέλεση αυτή τη στιγμή και για όλες τις πλευρές υπήρξε συμφωνία ότι τα προγράμματα είναι πολύ επιτυχημένα. Ε, το είπαν άλλωστε και οι ίδιοι. Ο επικεφαλής αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ικαράγουα και στον Παναμά και ο πρέσβης της ΕΚΑ, ο κ. Κένι Μπέλ, μας ενημέρωσε επίσης για τις νέες πολιτικές συνεργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ένα θέμα το οποίο ανέφερα πολλές φορές είναι κάτι που έχει και θετικά και αρνητικά. Τι εννοώ, ότι οι χώρες ε, μεσαίων εισοδημάτων όπως είναι ο Παναμάς και η Κωνσταντίνα δεν είναι επιλέξιμες για την ε, παραδοσιακή αναπτυξιακή βοήθεια. Απ' τη μια είναι θετικό το ότι αναπτύσσονται και έχουν ε, καλύτερα αποτελέσματα, αλλά το αρνητικό είναι ότι δεν θα μπορούν να λαμβάνουν τέτοιες ενισχύσεις. Αυτό το οποίο βέβαια διευκρινίστηκε σαφώ και μα εξήγησαν είναι ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μέσων συνεργασία και κυρίω ε, μέσα συγχρηματοδότησης με νέα μοντέλα πέραν της τεχνικής συνδρομής και της ε, τριμερού συνεργασίας. Επειδή θεωρούνται αυτές οι χώρες πλέον χώρες μεσαίου εισοδήματο, μπορούν να εποφοληθούν ε, αυτών των προγραμμάτων και της τριγωνικής συνεργασίας, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό. Όσον αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντρικής Αμερικής, ε, η γραμματεία της ε, ε, οικονομικής ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής της ΣΥΕΚΑ μας έδωσε ε, μια εικόνα της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Ε, εφαρμόστηκαν ή θα εφαρμοστούν σύντομα συγκεκριμένες νομοθεσίες, κυρίως όσον αφορά το σεβασμό των τελωνιακών και δασμολογικών νόμων και επίσης έχουν συσταθεί νέες αρχές που έχουν κοινή τελωνιακή εξουσία. Από την έναρξη ισχύω τη συμφωνία Σύνδεσης, ο όγκο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντρικής Αμερικής παρουσιάζει αύξηση και οι εξαγωγές Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κεντρική Αμερική αυξάνονται περισσότερο και αυξάνονται από σε σχέση με τις ε, εξαγωγές ε, της Κεντρικής Αμερικής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, από τη μία κατεύθυνση έχουμε πολύ ε, μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι από την άλλη. Και βάσει των όσων συζητήσαμε, υπήρξε μια συμφωνία να παρακολουθήσουμε το θέμα στενά, διότι όλοι σαφέστατα θέλουμε να λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτή η συμφωνία. Όσον αφορά το θέμα το οποίο συζητήθηκε περισσότερο και έλεγε και η Πρόεδρος ότι εδώ και τέσσερα χρόνια συζητιέται το θέμα της μελλοντικής ε, μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε πολύ μεγάλο διάστημα και ε, η Συμφωνία Σύνδεσης υπεγράφει το 2012 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κύρωσε στις 11 Δεκεμβρίου του 2012. Δηλαδή έχει περάσει πολύ καιρό. Είναι αλήθεια ότι οι χώρε τη Κεντρική Αμερική ε, στο μεταξύ κύρωσαν και αυτοί εδώ και πέντε χρόνια, το 2013 τη συμφωνία, αλλά υπάρχουν τέσσερις χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση που ακόμα δεν έχουν κυρώσει. Ε, θα πούμε ότι είναι τρει, γιατί έχουμε Αυστρία, Βέλγιο και Ελλάδα, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο ακόμα δεν έχει υπογράψει μένα, αλλά με τον Brexit νομίζω ότι δεν χρειάζεται και υπογραφή του. Ε, εκμεταλλεύουμε λοιπόν και την ευκαιρία αυτό που κάνουμε πάντα και το κάνει πάντα η Πρόεδρος ε, να προσπαθήσουμε να πείσουμε και αυτούς που δεν έχουν κυρώσει να κυρώσουν επιτέλους αυτή τη Συμφωνία Σύνδεσης. Η ίδια Συμφωνία Σύνδεσης ε, στο άρθρο 9 προέβλεπε ότι θα υπάρχει μια κοινή ε, μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή. από τη μια θα αποτελείται από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από την άλλη ε, μέλη του Παρλαθέν και ε, εκπροσώπους χωρών που δεν συμμετέχουν στο Παρλαθέν όπως για παράδειγμα έχουμε η Κωνσταντίνα. Η συζήτηση ε, οδήγησε σε ένα πρώτο σχέδιο κειμένου το 2014 και υπήρξε συμφωνία για ένα κανονισμό. Εκεί προτάθηκαν να υπάρχουν 15 μέλη που είναι η συνήθι σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από την άλλη πλευρά μέλη του Παρλασέν και μέλη της ε, συνέλευσης της Κωνσταντίνας ε, και θα είχαν και αυτοί 15 μέλη. Εμείς ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2015 εγκρίναμε αυτό τον κανονισμό και επομένω είμαστε σωστοί, αλλά με μία επιστολή ε, της 29 ε, 29 Μαρτίου του 2017 η νομοθετική συνέλευση της Κώστα Ρίκα εξέφρασε την διαφωνία της για την πρόταση του Παλαιστέν όσον αφορά τη σύνθεση και τον αριθμό των μελών της Επιτροπής και ζήτησε αντί για 15 μέλη για κάθε πλευρά να έχει 12 μέλη κάθε πλευρά. Εμείς ε, συνεχίσαμε να θέτουμε το θέμα και λέμε ότι θα πρέπει να παραμείνουν τα 15 μέλη. Η Κωνσταντίνα ισχυρίζεται ότι πρέπει να είναι 12, 12-2 ε, για κάθε μία από τις χώρες ε, της ε, Παρλασέν και το θέμα περιπλέκεται γιατί θα πρέπει να δώσουμε εδώ και τη δυνατότητα στη Δομινικανή Δημοκρατία, η οποία πρέπει να συμμετέχει σε αυτή την επιτροπή, δεδομένου ότι είναι μέλος του Παρλασέν και του ΣΥΚΑ παρά το γεγονός ότι δεν ε, αποτελεί τμήμα της Συμφωνίας Σύνδεσης. Εδώ λοιπόν περικλέκονται λίγο περισσότερο τα πράγματα. από τη μια ε, αυτοί που ε, δεν είναι μέλη του Παρλασέν και πρέπει να συμμετέχουν όπως η Κωνσταντίνα και αυτοί που είναι μέλη του Παρλασέν ε, και δεν έχουν συμφωνία όπως είναι η Δομινικανή Δημοκρατία. Μία λύση που προτάθηκε θα μπορούσε να είναι η Δομινικανή Δημοκρατία να συμμετέχει ως παρατηρητής. Ε, πιστεύουμε ότι είναι ευπρόσδεκτοι και πρέπει να συμπεριληφθούν και ότι σε αυτό το καταμερισμό των 15 μελών θα πρέπει να συμφωνήσουν πώς θα ε, μοιραστούν μεταξύ των έξι χωρών συν τη Ρίκα και τη Δομανικανή Δημοκρατία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε συνέχεια το θέμα. Πρέπει να βρεθούμε μια λύση. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε πρέπει να βρεθεί μια λύση και Έχουμε προβλέψει να γίνει και μία συνεδρίαση πριν από τη Γιούρελά του Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Και στη συνεδρίαση της Eurolat του Σεπτεμβρίου του 2018 να υπάρξει μια κοινή πρόταση οριστική και να έχει υπάρξει και συμφωνία από αυτού. Αυτή είναι η διάθεση που υπάρχει. Αλλά εάν πραγματικά θέλουμε να υπάρξει συμφωνία το Σεπτέμβριο του 2018, θα πρέπει να υπάρξει και μια κοινή πρόταση μεταξύ Παρλασέν, Κώστα Ρίκας και Δομινικανής Δημοκρατίας, γιατί εμείς ε, υπ' αυτού του όρου τη σύνθεση 15-15 δεν σκοπεύουμε να παρεύουμε και θα σεβαστούμε απολύτω τη θέση ε, που έχετε εσείς για την κατανομή των 15 ε, μελών. Τίποτα άλλο, αν έχετε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Νομίζω ότι σας έδωσα πλήρως πληροφορίες για το τι συνέβη. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Η ενημέρωση ήταν πλήρης. Ε, όσον αφορά την πρόοδο της Συμφωνίας Σύνδεσης. Θα σταθώ στο τελευταίο που είπατε για τη Συμφωνία να εκπονηθεί κοινή ε, ε, πρόταση για τον ιστορικό κανονισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Παρλασέν, Κωνσταντίνα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από τη συνεδρία των τριών μερών, με την ελπίδα ότι και οι τρεις χώρες που απομένουν θα υπογράψουν τη Συμφωνία Σύνδεσης ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίε ε, και να προχωρήσει η συμφωνία σε όλο τη το έβρο. Τώρα να πάμε στο πέμπτο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορούν στις βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Φεβρουαρίου και την 1η Απριλίου του 2018 στην Κωνσταντίνα για την εκλογή νέου Προέδρου και νομοθετικής συνέλευσης και να σας πω ότι συγκεκριμένα στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου μεταξύ του κυρίου Μουνιώθ από το Συντηρητικό Κόμμα της Εθνικής Αποκατάστασης που εξασφάλισε το 24% των ψήφων και του συγγραφέα και πρώην Υπουργού Κάρλος Κεσάδα από το Προοδευτικό Κόμμα Δράση των Πολιτών που απέσπασε το 21% των ψήφων, ε, με δεδομένο ότι κανένα υποψήφιο δεν έλαβε κατά την ψηφοφορία του πρώτου γύρου που πραγματοποιήθηκε στην 1η Απριλίου του 2018 περισσότερο από το 40% των ψήφων, η χώρα πήγε σε δεύτερη εκλογική διαδικασία, στην οποία επικράτησε ο κ. Κεσάδα με 60,8% των ψήφων. Πρέπει να πούμε ότι η προεκλογική εκστρατεία έλαβε έντονα χαρακτηριστικά αντιπαράθεση έπειτα από την απόφαση τη 9η Ιανουαρίου του 2018 του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οποία η Κώστα Ρίκα πρέπει να νομιμοποιήσει τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, μια απόφαση με θεωρητικό επίπεδο, που σε θεωρητικό επίπεδο δεσμεύει ω προ την εφαρμογή τη ολόκληρη την Λατινική Αμερική και ω εκ τούτου η προεκλογική εκστρατεία συμμαδέστηκε από την έντονη αντιπαράθεση για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, με τον πρώτο γύρο να παίρνει διαστάσει δημοψηφίσματο για το ακαθόδε αυτό ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο υποψήφοι για το αξίωμα του Προέδρου έλαβαν προεκλογικά και διαμέτρου αντίθετε θέσει επί του θέματο. Ο κ. Μουνιώθ, που πριν την έκδοση τη απόφαση του δικαστηρίου φερόταν να εξασφαλίζει τη βάση των δημοσκοπήσεων γύρω στο 3%, διεξήγαγε μια εξαιρετικά επιθετική εκστρατεία κατά τη νομιμοποίηση των γάμων μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών και κατόρθωσε να πάρει την πρώτη θέση στι προεδρικέ εκλογέ του πρώτου γύρου στι 4 Φεβρουαρίου. Αξίζει επίση να σημειωθεί ότι οι δημοσκοπήσει προέβλεπαν αμφίροπη μάχη, ωστόσο η έκβαση τη αναμέτρηση αποδείχθηκε θεματικά διαφορετική, καθότι ο κύριο Κεσάδε επικράτησε στο δεύτερο γύρο με διαφορά περίπου 20 μονάδων. Επιπλέον, η ψηφοφορία για την νομοθετική συνέλευση προκάλεσε τον παραπέρα κατακαιρματισμό του πολιτικού σκηνικού στη χώρα το Κόμμα Εθνικής Απελευθέρωσης κέρδισε 17 έδρες, το Εθνικό Κόμμα αποκατάσταση κέρδισε 14 έδρες, το Κόμμα δράση των Πολιτών κέρδισε 10 έδρες, το Κόμμα κοινωνική χριστιανική ενότητα κέρδισε 9 έδρες, το Εθνικό Κόμμα ένταξη κέρδισε 4 έδρες, κέρδισε 2 έδρες και το αριστερό ευρύ μέτωπο και το ε, ε, ευρύ αριστερό μέτωπο κέρδισε 1 έδρα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να μου επιτρέψετε να δώσω τον λόγο στην αυτή εξοχότητα των πρέσβη της ε, Κωνσταντίνα, τον κύριο, κύριο Αλφάρο, για να μας ε, σχολιάσει τη διενέργεια των εκλογών στη χώρα του. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Μάτο, αξιότιμοι βουλευτές και συνάδελφοι πρέσβης και διπλωμάτες που μας συνοδεύουν, κύριοι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Γραμματείας της Αντιπροσωπείας, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που σας ε, χαιρετίζω εδώ, ε, δεχόμενος την πρόσκληση της ε, αντιπροσωπείας των χωρών της Κεντρικής Αμερικής για να μπορέσω να σας κάνω μια παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εκλογών. Στις 4 Φεβρουαρίου και στη 1 Φεβρουαρίου οι κάτοικοι της Κώστα Ρίκας προσέφηγαν στις κάλπες ε, και είχαμε κληθεί να λάβουμε μια απόφαση για όλη τη χώρα, να επιλέξουμε τους ε, κυβερνήτες μας για το διάστημα 2018-2022 που θα είναι η κυβέρνηση ε, της επαιτίου και των 200 ετών ε, της ίδρυσης της χώρας μας. Και επίσης θα ήθελα να σας πω και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία αυτών των εκλογών. Καταρχάς, Το εκλογικό σώμα ήταν κάτι παραπάνω από 3 εκατομμύρια. Μας ε, ζητήθηκε να ασκήσουμε τα εκλογικά μας δικαιώματα και να επιλέξουμε μεταξύ τριών υποψηφίων για την Προεδρία της Δημοκρατίας, δύο αντιπροέδρων και 56 ε, μέλη ε, της Βουλής για την επόμενη θητεία. Επίσης, εκλογικό σώμα κατά 50%, 50,18% αποτελούνταν από γυναίκες και 49,82% από άντρες. Από το συνόλο του εκλογικού σώματος το 50% ήταν μεταξύ 18 και 40 ετών. Είχαμε πάνω από 61.000 άτομα τα οποία είχαν λάβει ηθαγένεια Κωνσταντίνα που μπορούσαν να ψηφίσουν, πάνω από 36.000 άτομα τα οποία ανήκαν στις αυτόχθονες ε, κοινότητες των διαφόρων περιοχών ε, και υπήρξε μετάφραση λοιπόν και στις πέντε γλώσσες των αυτοχθόνων και υπήρχαν και ε, 1.575 άτομα τα οποία ψήφισαν ε, σε διάφορα εκλογικά κέντρα στις φυλακές. Και είχαμε τα εξή αποτελέσματα, δεν θα αναφέρω κάποιο από αυτά τα οποία είπε ήδη η Πρόεδρος. Ξεκινάμε από, την, ε, από το Εθνικό Κογκρέσο, τη Βουλή, είχαμε επιλογή των βουλευτών, οι βουλευτές και αναπληρωτές, ε, όλοι εκλέγονται για κάθε μία από τις 7 περιφέρειες βάσει και του πληθυσμού για την επόμενη περίοδο 2018-2022 έχουμε 7 κόμματα στη Βουλή τον αριθμό των βουλευτών τον ανέφερε η Πρόεδρος. Ε, θα αναλάβουν καθήκοντα από 1η Μαΐου και θα επιλέξουν και το Προεδρείο για το διάστημα 2018-2022 βάσει και των συνταγματικών ε, κανόνων που καθορίζουν ότι το Προεδρείο επιλέγεται κάθε χρόνο και όχι κάθε τέσσερα χρόνια. Ε, όσον αφορά τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, έγινε ένας πρώτος γύρος ο οποίος ε, ε, δεν θεωρείται πρώτος γύρος αν δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα για πρόεδρο και αντιπρόεδρο ε, στον οποίο ε, μόνο τέσσερα πολιτικά κόμματα πήραν από, πάνω από 10% των ψήφων. Είχαμε τρεις υποψηφίους, επομένως οι πολίτες είχαν αρκετές επιλογές. Αυτοί που έλαβαν πάνω από το 10% ήταν το αξιόν σου να δάναμε με πάνω από 25%, είχαμε ένα κόμμα με πάνω από 18% και το κόμμα χριστιανικής ενότητας ε, ε, πάνω από 16%. Όσον αφορά τη σύνθεση, επειδή κανένας από τους υποψηφίου δεν πήρε ε, το ποσοστό το οποίο προβλέπεται, η Εφορευτική Επιτροπή βρήκε μια λύση και κάλεσε για ένα δεύτερο γύρο με τους δύο υποψηφίους που είχαν λάβει τις περισσότερες ψήφους. Σε αυτό το δεύτερο γύρο το αποτέλεσμα ήταν να κερδίσει το κόμμα της δράσης των πολιτών με 60,59% των ψήφων και το δεύτερο κόμμα, της ε, ε, Εθνικό Κόμμα Αποκατάστασης, πήρε 39%. Ε, ε, εξελέγει λοιπόν ο κύριος Κάρλος Αλβαράδο Κεσάδα, ο οποίος θα είναι ο 58ος πρόεδρος ε, της Δημοκρατίας για το διάστημα 2018-2022. Να πω ότι η κυρία Εψή Κάμπελ Μπάρ θα είναι η πρώτη γυναίκα αφρικανικής καταγωγής που θα λάβει θέση αντιπρόεδρου στην Κωνσταντίνα και κατά πάσα πιθανότητα και στην υπηρετική Λατινική Αμερική. Και αυτό φυσικά συνάδει πλήρως με τις αξίες που έχουμε κοινέ με την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κωνσταντίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα την ε, ε ισότητα των φύλων. Η Κωνσταντίνα προωθεί την πραγματική πρόσβαση των γυναικών σε διευθυντικές ε, θέσεις και πολιτικές θέσεις, όπως για παράδειγμα ε, από το 1900 86 επιλέξαμε την πρώτη αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας και φέτο, ε, την ίδια χρονιά για πρώτη φορά μια γυναίκα προέδρευσε ε, στο Εθνικό Κογκρέσο. Πρόκειται λοιπόν για συγκεκριμένα γεγονότα και αυτά μας επιτρέπουν να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι από τις εκλογικές ε, λίστες στις οποίες είχαμε επικεφαλής γυναίκες το 2014 περάσαμε από το 22% στο 43% το 2018. Ο νέος πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του ναι, θα αναλάβουν καθήκοντα σε μια έκτακτη σύνοδο της ε, ε, Βουλής ε, στις 8 Μαΐου του 2018 και θα γίνει ορκομοσία του Προέδρου και των Αντιπροέδρων. Και μετά ο Πρόεδρος θα επιλέξει και το Υπουργικό του Συμβούλιο. Η Εφορευτική Επιτροπή έτσι ενισχύει τη θέση του ως βασικός ε, μοχλός ε, της ε, λειτουργίας της Δημοκρατίας της Κωνσταντίνα και αυτό φυσικά δεν θα πρέπει να το λησμονούμε. Είναι πυλώνας και αποτελεί την τέταρτη εξουσία της Δημοκρατίας με ανεξαρτησία και υψηλό τεχνικό επίπεδο. Ανεξαρτησία η οποία παρέχεται βάσει του συντάγματος. Ως τμήμα των εργασιών της και με τη στήριξη της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών έγινε μια εκστρατεία που καλούσε τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν για να μειώσουμε την αποχή, κάτι το οποίο επετεύθη στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Επιπλέον, αυτή η εκλογική διαδικασία ε, είχε και αρκετούς παρατηρητές, ε, τους οποίους είχε καλέσει η Εφορευτική Επιτροπή και ε, η Υπήρχε και ε, παρατήρηση των εκλογών από τις αμερικανικές ε, χώρες και είδαμε ότι υπήρχε πνεύμα συνεργασίας ε, και πριτάνευσε αυτό μεταξύ των διαφέρων φορέων καθώς επίσης και την ίδια ημέρα, την ημέρα των εκλογών. Η αποστολή που ανέλαβε ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας, ο Αντρές Παστράνα, ε, χαιρέτησε με τον επαγγελματισμό με τον οποίο διοργανώθηκαν αυτές οι εκλογές ε, και ανέφερε και μια σειρά από καλές πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν και σημείο αναφορές για άλλες χώρες της περιοχής. Και αναφέρω μεταξύ αυτών ε, τις πρωτοβουλίες ε, του ε, εκλογικού δικαστηρίου για να μπορούν να ψηφίσουν ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία, το να υπάρχουν οθόνες ψηφοφορίας και να υπάρχουν και δυνατότητες για να μπορέσουν να προσφέρουμε στους πολίτες πληροφορίες για την εκλογική διαδικασία. Η αποστολή ε, παρατηρητών των εκλογών ε, τόνισε ότι υπήρχε μεγάλη εκλογική επάρκεια και επίσης ε, έγιναν αρκετές συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης. Ε, υπενθύμησε τη συζήτηση για το σύστημα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και επίσης συζητήθηκαν και θέματα ισότητας. Και στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο Τονίζεται η ταχύτητα με την οποία έγινε επεξεργασία των δεδομένων που επέτρεψε να έχουμε αποτελέσματα σε πολύ λίγες ώρες μετά από την ώρα που έκλεισαν οι κάλπες. Ε, το ανώτατο εφερευτικό δικαστήριο ανακοίνωσε και τα τελικά αποτελέσματα, όπως γίνεται συνήθως, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό μετά από μια εκστρατεία η οποία ε, χαρακτηρίστηκε από πόλωση της κοινωνίας, όπως για παράδειγμα ο γάμος των ομοφύλων ζευγαριών ε, και ε, θέματα μαθημάτων σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία. Ε, και οι δύο υποψήφοι με πολύ πολιτισμένο πλεύμο ε, χαιρετήθηκαν και ο καθένας αναγνώρισε φυσικά τα αποτελέσματα των εκλογών. Όπως βλέπετε πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο σίγουρα μπορεί να τελειοποιηθεί. Έχει κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις οι οποίες εξακολουθούν να εμένουν αλλά και οι δύο υποψήφοι ε, σε αυτό το δεύτερο γύρο ήξεραν ότι Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι προγραμματικοί στόχοι και αυτό προσπαθεί να κάνει από εδώ και πέρα ο νικητή. Γι' αυτό όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας, η Κωνσταντίνα θα συνεχίσει να εργάζεται προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει ε, να... Ε, εξετάζει το θέμα και να αναθεωρήσει και να μην υπάρχει διαίρεση μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, αλλά να είμαστε μία περιφέρεια και να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την συνεργασία, η οποία είναι απαραίτητη, διότι υπάρχουν ε, προκλήσεις. Κυρίες και κύριοι, ως μία από τις πιο μακροχρόνιες και σταθερές δημοκρατίες της Λατινικής Αμερικής και της Κεντρικής Αμερικής, η συμμετοχή στις εκλογές για τους κατοίκους της Κωνσταντίνας είναι μία συνάντηση με τις ρίζες τους ο καφές μας, η βιοποκυλότητά μα και η υψηλή τεχνολογία μεταξύ άλλων είναι αυτοί που μας διακρίνουν ε, ανά τον κόσμο. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο παρά η δημοκρατική μας ε, παράδοση. Εμείς οργανώνουμε τη ζωή, σας, τη ζωή μας από κοινού με ειρήνη και ελευθερία. Η Κωνσταντίνα σήμερα μπορεί να παρουσιάζεται στον κόσμο αλλά και στην ίδια τη χώρα που ως μια διαδικασία τακτική, ε, μια συμμετοχική διαδικασία που επιτρέπει να έχουμε ένα ε, σύστημα πολυφωνίας που σέβεται το κράτος δικαίου και έχει και κοινωνικό όραμα, είναι τους πάντες πολυεθνικό και πολυπολιτισμικό. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για αυτά τα αποτελέσματα και ελπίζουμε να μπορέσουμε να εργαζόμαστε συνεχώς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτή την αντιπροσωπεία και με όλα τα ε, σχετικά όργανα και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Ευχαριστώ μία ακόμα φορά, Πρόεδρε καταρχήν να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να συγχαρώ τον ε, πρέσβη για τα εκλογικά αποτελέσματα και κυρίως ε, τον κύριο Κάλβος Κάρλος Αλβαράδο που εξελέγει πρόεδρος της Κωνσταντίνα. Του ευχόμαστε στον ίδιο και στην κυβέρνησή του καλή επιτυχία και την ευκαιρία να συγχαρώ την Κώστα Ρίκα για τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η εκλογική διαδικασία, για την ταχύτητα στην καταμέτρηση, την υψηλή συμμετοχή του εκλογικού σώματος και οπωσδήποτε και για το αποτέλεσμα το οποίο είναι σαφές και δεν αφήνει περιθώρια παρεμηνιών. Θα επιτρέψει στον πρόεδρο Αλβαράδου να συνεχίσει το θετικό του ε, και προοδευτικό έργο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κωνσταντίνα έχουν εξαιρετικέ διμερεί σχέσει. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά και στο διεθνέ περιβάλλον, πολυμερό. Θέλουμε να συνεχίσουμε και να εμβαθύνουμε αυτή τη συνεργασία στο μέλλον κατά τη διάρκεια τη επόμενη θητεία. Επί τη βάση κοινών αρχών θα ενισχύσουμε την ήδη στενή συνεργασία μας και επίσης ε, προασπίζοντας ε, κοινέ ε, αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο πολυμερού συνεργασίας που γίνεται όλο και πιο σημαντική, πιο σημαντική από ποτέ προκειμένου να προασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμού την, κατα... την, κατα... την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την προασπίση του περιβάλλοντος προκειμένου οι κοινωνίες μας να είναι όλο και πιο ευημερούσες χωρίς αποκλεισμού. Κωνσταντίνα αντιμετωπίζει βέβαια προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει στο πλευρό της ε, για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και για να προχωρήσουμε όπως σε θέματα όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς, η ασφάλεια των πολιτών που είναι και περιφερειακό και παγκόσμιο πρόβλημα και βέβαια τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, οι κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις στις οποίες αναφέρθηκε και ο πρέσβης. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, είναι πολύ προσιλωμένη στη συνεργασία της συνολικά με την Κεντρική Αμερική, όπως και η ε, Κωνσταντίνα, ε, που στο πλαίσιο του ΣΥΚΑ, το ΣΥΚΑ, αυτός ο, ο μηχανισμός ολοκλήρωσης Κεντρικής Αμερικής, απαιτεί την συνένεση όλων των μερών του και Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ε, Κώστα Ρίκα που ε, είναι και αυτή προσιλωμένη σε αυτό το περιφερειακό ε, σχέδιο ολοκλήρωσης. Η συμφωνία σύνδεσης, για παράδειγμα, είναι εξαιρετικά φιλόδοξη. Εδώ και αρκετό καιρό Έχουμε αυτή τη συνεργασία με όλη την Κεντρική Αμερική, αλλά επίσης και η Συμφωνία Πολιτικής Συνεργασίας και Διαλόγου, που μας ε, επιτρέπει να σημειώσουμε μεγάλη πρόοδο, να συναντιόμαστε, να αποφασίζουμε κοινή δράση. Είναι απόλυτα σημαντικό προκειμένου να υποφελούμαστε ε, στο μέγιστο δυνατό βαθμό των δυνατοτήτων που μας δίνονται. Άλλη μια φορά λοιπόν σας συγχαίρω για αυτή τη διαδικασία, για αυτό το αποτέλεσμα και εύχομαι στον πρόεδρό σας καλή επιτυχία. Το λόγο έχει ζητήσει ο συνάδελφος ο θα προσπαθήσω να μιλήσω μισά πρωτοβαλικά, μισά ισπανικά. Ε, δύο λόγια μόνο, γιατί θέλω και εγώ να συγχαρώ τον πρέσβη κύριο Άλβαρο για τον τρόπο με τον οποίο συμμετείχε ο λαός της Κωνσταντίνα ε, σε αυτές τις εκλογές. Τόσο το εκλογικό σώμα όσο και η αρχές ε, έπραξαν άριστα, δεν είναι κάτι καινούριο για μας, είναι παραδοσιακό στην Κωνσταντίνα, συγχαρητήρια και χαιρετισμού. Ε, είσαστε ένα πολύ καλό παράδειγμα δημοκρατία στην Λατινική Αμερική. Συγχαρητήρια. Αν και είναι μόνο για λόγους ευγένειας μετά από τις εξηγήσεις που μας έδωσε ο πρέσβης, δεν έχω πολλά να προσθέσω, να σας συγχαρώ και να σε ευχηθώ κάθε επιτυχία και όπως πάντα γνωρίζετε ότι εδώ έχετε φίλους ε, και πολιτικά αλλά και προσωπικά. Εγώ ε, ε, θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κοινοί δεσμοί ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ τον κύριο Πρέσβη, ευχαριστώ τους αδέλφους. Καλή επιτυχία κύριε Πρέσβη. Έχουν γίνει εκλογέ και στο Ελσαλβαδόρ, αλλά δεν μπορούσαμε να, κάνουμε συζήτηση σήμερα ακριβώ γιατί η Λίλια πρέσβη, οπότε μα ήταν αδύνατο να γίνει αυτό. Να ρωτήσω στου συναδέλφου αν έχουν κάποια άλλα θέματα να θέσουν. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Bueno. <clears throat> Señora Presidente, yo tengo... Ε, σας ε, σέβομαι πάρα πολύ, το ξέρετε πολύ καλά πρόεδρε, είμαι πάντοτε παρόν. Προσπαθώ να είμαι πάντοτε εδώ, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι συναντήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τις χώρες Κεντρικής Αμερικής. Αλλά ε, δεν είναι όλα ρόδινα. Πιστεύω ότι αυτή η αντιπροσωπεία δεν μπορεί να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορούμε αφενός να κλέμε για το θάνατο ενός δικτάτορα. Προφανώς μιλώ για τον Φιντελ Κάστρο. Ή αν το κάνουμε θα πρέπει να κλέμε και για τα θύματα του καθεστώτος. Αλλά κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι αυτή η αντιπροσωπεία δεν μπορεί να αγνοήσει την τραγωδία που ζουν οι αντιπολιτευόμενοι των δικτατόρων. Κοιτάξτε τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ικαράγουα με την τρομακτική βία η καταστολή του δικτατορικού καθεστώτος των Σαντινίστας. Αυτό δεν είναι ε, αποδεκτό. Νόμιζα ότι θα είχαμε ε, ένα ζήτημα στην μέση διάταξη για να συζητήσουμε για τα αυτά που έγιναν στην Ικαράγουα αλλά και στην Κούβα. Και θα σας πω τι νομίζω ότι έχει λάβει χώρα στην Κούβα, αλλά στην Ικαράγουα ε, ο πρόεδρος του των Σαντινίστας ε, ε, προσπάθησε να επιβάλλει κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες προκάλεσαν 30 ε, θανάτους, 428 τραυματισμένους ε, και πάρα πολλούς φυλακισμένους και εξαφανισμένους που σημαίνει συχνά εκεί. Δεν μπορούμε να σιωπήσουμε χωρίς ε, να καταδικάσουμε επίσημα με την αποστολή επιστολής ε, στην πρεσβεία της Νικαράγουας στις ε, Βρυξέλλες καταδικάζοντας λέω την καταστολή του λαού της Νικαράγουας. Επίσης δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι έναντι της καταστολής τρεις μέρες μετά την ε, ε, ε, εκλογή του νέου πρόεδρου της Κούβας εναντίον των Ντάμας Εμπλάνκο που γνωρίζετε έχουν κερδίσει και το βραβείο Νόμπελ. Πιστεύω ότι η αντιπροσωπεία μας πρέπει να αποστείλει επιστολή και στην πρεσβεία της Κούβας ε, ε, καταδικάζοντας την αφαίρετη φυλάκιση των δύο γυναικών και να ζητάμε την απελευθέρωσή τους. Πέραν από τις ε, επιστολές συγχαρητηρίων ε, μετά από δίθεν δημοκρατικές εκλογές, μετά από μια δίθεν δημοκρατική εκλογή ε, και ξέρουμε ότι ήταν μια φάρσα γιατί έγιναν δια, διαμαρτυρίες και αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό, ε, θα πρέπει να εκφράσουμε την ε, αντίθεσή μας με αυτό το καθεστώς και με αυτή την κυβέρνηση της Κούβας. Και εγώ και άλλοι συνάδελφοι πιστεύουμε ότι αυτή θα πρέπει να είναι η δράση μας έναντι των δύο ε, πρεσβειών. Ε, δεν είναι δυνατόν να έχουμε τις, τα τόσα καλά παραδείγματα της Κώστα Ρίκα, του, του Ελσαλβαδόρ και άλλων χωρών της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής ε, και να έχουμε ταυτόχρονα αυτούς τους λεκέδες της δημοκρατίας, τους λεκέδες πάνω στη δημοκρατία ε, όπως αυτές οι δύο χώρες, ε, Νικαράγουα και Κούβα. Η καταστολή ε, στην Κούβα είναι απαράδεκτη. Ο κύριος ε, πρέσβης της Κωνσταντίνας μίλησε για τις κοινέ μας αξίες με, την, ε, με τις χώρες Κεντρικής Αμερικής ε, αλλά όχι όλες τις χώρες Κεντρικής Αμερικής κύριε Άλβαρο γιατί στη δική σας περιοχή υπάρχουν χώρες που δεν είναι δημοκρατικές και που δεν προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να καταδικαστούν κύριε Πρόεδρε αυτές οι αντιλήψεις και οι καταστολή τόσο στην Ικαράγουα όσο και στην Κούβα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε και πρέπει να εξηγήσω κάποια πράγματα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Καταρχήν, στο σημείο 2 της ε, μερίσιας διάταξης αναφέρθηκα εκτενώς σε ό,τι έγινε στην ε, Νικαράγουα και στους 30 θανάτους και πολύ σωστά ο κύριος Μάτο παρατήρησε και αποδέχθηκα να κάνουμε κάποια επιστολή. Αυτό θέλω να το ξέρετε, δεν ήσασταν παρόν εκείνη τη στιγμή. Όσον αφορά τώρα το θέμα της Κούβας. Καταρχήν θεωρώ ότι από τη θέση μου δεν μπορώ να χαρακτηρίσω απολύτως τίποτα και δεν έχω πάρει μέρος είτε αν στηρίζω ή δεν στηρίζω. Πρέπει η θέση μου να είναι ουδέτερη και αυτό προσπαθώ να κάνω όσο καιρό βρίσκομαι σε αυτή την έδρα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε μια σύναψη συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κούβα. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Είμαι υποχρεωμένη λοιπόν και πάλι από τη θέση μου να κρατήσω μια τυπική διαδικασία και σε έναν εκλεγμένο από εκείνους πρόεδρο να στείλω μια συγχαρητήρια επιστολή. Τυπική συγχαρητήρια επιστολή που θέλω να πιστεύω ότι δεν παίρνει μέρος, δεν εκφράζει πολιτική άποψη, είναι μια τυπική επιστολή συγχαρητηρίων. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε. Ο κύριο Μάτο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι στο σημείο 2 η πρόεδρος αναφέρθηκε στην Νικαράγουα και εγώ είπα σαφέστατα ότι πρέπει να πούμε την άποψή μα και συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε ο συνάδελφο Φαρία γιατί υπάρχει ταύτιση απόψεων. Και εγώ είπα σαφέστατα στην πρόεδρο ότι όπως ε, ε, στείλαμε τα συλληπιτήριά μας και συγχαρήκαμε στη συνέχεια πρέπει να καταδικάσουμε και την ε, καταστολή ε, στην Ικαράγουα και φυσικά θα πρέπει να στείλουμε και μια πολύ αυστηρή επιστολή το επαναλαμβάνω γιατί δεν ήσασταν εδώ δεν ήταν και ο πρέσβης της Νικαράγουας ε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι καταδικάζουμε ακράδαντα αυτή την ε, ε, βάναυση ε, καταστολή και την αλληλεγγύη μας προς τα θύματα και τους τραυματισμένους. Το ξαναλέω, δεν ξέρω αν ήταν ή αν δεν ήταν, αλλά το είπα σαφέστατα και η Πρόεδρος είπε ότι αυτό θα κάνουμε. Ε, τίποτα άλλο, δεν έχω κάτι να επαναλάβω, συμφωνώ με τα όσα είπε ο κ. Φαρία, ε, ο οποίος δεν με είχε ακούσει, αλλά εγώ τον άκουσα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, για άλλη μια φορά να σας πω ότι σας εκτιμώ ιδιαίτερος. Εκτιμώ ιδιαίτερος τη στάση σας και πιστεύω ότι εσείς ε, εκπροσωπείτε πολύ καλά την αντιπροσωπεία. Δεν είπα τίποτα το αντίθετο, να μην παρεξηγήσετε. Αλλά πιστεύω ότι όταν ανακύπτει ένα τέτοιο θέμα, τέτοιες καταστολής, ε, εμείς περιμένουμε από εσά ως αντιπροσωπεία να ε, ε, δράσετε γιατί είναι επίγον το θέμα. Δεν ήμουνα, ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν από την αρχή, το ξέρετε όμως ότι τρέχουμε από τη μία συνεδρία στην άλλη. Είμαι εδώ γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που μιλήσετε γι' αυτό και να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Γκαμπριελ Μάτο που ε, δήλωσατε τη συγκεκριμένη πρόθεση. Αλλά εσείς κυρία Πρόεδρε είπατε κάτι με το οποίο διαφωνώ. Ε, γιατί εκλογές μιλάτε, τι εκλογή εννοείτε. Αναφέρεστε σε εκλογές, αλλά εγώ δεν γνωρίζω να συνέβη κάποια εκλογή. Ναι, είχαμε εκλογές στην Κωνσταντίνα, ναι, στην Παραγουάη, έχει πολλές, αλλά στην Κούβα ε, δεν άκουσα να διεξάγονται εκλογές. είχαμε το αποτέλεσμα χωρίς εκλογή και το οποίο οδήγησε σε διαδηλώσεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τραυματίες και ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φυλακή. Η Ντάμας Ντεμπλάνκο που έλαβαν βραβείο Ζαχάροφ το 2015. Και κάτι άλλο κυρία Πρόεδρε που ξέχασα. Η αντιπροσωπεία μας θα πρέπει να ζητήσει από τις αρχές της Κούβας να μην απαγορεύσουν στους ε, νικητές του κερδίου του βραβείου για την ελευθερία ε, να πάνε στις 17 Μαΐου στη Νέα Υόρκη για να λάβουν το βραβείο. Ε, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια διαμαρτυρία, απλώ ε, θα πάνε για να βραβευθούν. Νομίζω ότι αυτή τη στάση πρέπει να τηρήσει η αντιπροσωπεία μα, κυρία Πρόεδρε. Σαφώ, κυρία Πρόεδρε, εσεί πρέπει να βρίσκεστε υπεράνω άλλων και να είστε ανεξάρτητοι και σα ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτή είναι η στάση σα. Αλλά όχι η δική μου. Εγώ πρέπει να καταδικάζω τα πράγματα ω έχουν. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Ε, ευχαριστώ. Για να κλείσουμε με αυτό το θέμα και υπό το φω των όσων ακούγονται, ε, θα ήθελα επισήμω να σα ζητήσω στην επόμενη συνεδρίασή μα να γίνει μια συζήτηση για την Ικαράγουα. Αν πρέπει να το συμφωνήσουμε, ας το συμφωνήσουμε επίσημα, καλώντας βέβαια και τον πρέσβη για να συμμετάσχει. Είχα και άλλο θέμα, αλλά ίσω ο κ. Φαρία θέλει να προσθέσει κάτι. Ε, έχω κάποιο άλλο θέμα άσχετο με αυτό. Και άλλη μια πρόταση για την αντιπροσωπεία μα: ε, ε, να έχετε ένα ξυπνητήρι για να μην αποκοιμούνται οι άνθρωποι. Τελευταίο δεν τα άκουσα κύριε Φαρία. θα με επιτρέψετε και πάλι να πω ότι στάση μου, πολιτική μου είναι να μην μπαίνω σε εσωτερικέ διαδικασίε καμιά χώρα και ειδικά όσον αφορούν εκλογέ. Αυτό, από αυτή τη θέση που βρίσκομαι, κάτω από αυτό το έδρανο μπορώ να, να έχω άποψη και μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση ανοιχτή και οι δύο. Βεβαίω και θα κάνουμε τη συζήτηση που, που είπατε. Μπορούμε να δεσμευτούμε σε αυτή την αίθουσα τώρα, στην επόμενη συνεδρίαση, η οποία θα γίνει, όπω πολύ καλά ξέρετε, στι 28 Ιουνίου του 2018 εδώ στι Βρυξέλλε. Εάν δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, λίγη συνεδρία. Ευχαριστώ όλους τους κυρίους και τις κυρίες που βρίσκονται σήμερα εδώ στην... Έχω και κάτι ακόμα. Ε, πιο ειρηνικό, κυρία Πρόεδρε, για τις ε, αντιπροσωπείες της ε, τι αποστολέ μάλλον τη αντιπροσωπεία μα. Την τελευταία χρειάστηκε να την ακυρώσουμε γιατί δεν υπήρχε ανεπαρκή αριθμό μελών, αλλά νομίζω ότι τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να πάμε στη Γουατεμάλα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και ελπίζω ότι ο πρέσβης θα το δεχτεί με ικανοποίηση. Πιστεύω ότι η Γουατεμάλα πληρεί όλε τι προποθέσει ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να ε, ε, το επισκεφθεί και να έχουμε μια αποστολή της αντιπροσωπείας μας. Ε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα τέτοιο ταξίδι. Έχουμε προβλέψει και την Κούβα, αλλά πάντα προβλέπουμε την Κούβα και τελικά δεν μπορούμε να πάμε. Ε, εκτός και αν μας αφήσουν να πάνε με απόλυτα ελεύθερο πρόγραμμα από πλευράς μας. Επειδή δεν θα συμβεί λοιπόν κάτι τέτοιο, νομίζω ότι αντί να περιμένουμε συνεχώς ε, την πρόσκληση, καλό είναι να πηγαίνουμε σε χώρες φίλους που μας περιμένουν και μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα εκεί. Ε, και συγγνώμη και κάτι ακόμα που το ε, αναφέρατε κυρία Πρόεδρε, το Ελσαλβαδόρ. Ξέρω ότι θα το συμπεριλάβατε στην επόμενη συνεδρίαση, αλλά μου είπε ότι ο επικεφαλής της ε, αποστολής παρατήρησης ότι πολύ θα χαιρόταν να έρθει εδώ και να εξηγήσει και ε, ξέχασα να το πω όταν είπατε για το Ελσαλβαδόρ, ότι πολύ ευχαρίστως ε, θα ήθελε να έρθει εδώ. Άρα λοιπόν στην επόμενη συνεδρίαση, στην ημερήσια διάταξη, θα έχουμε ως θέμα το Ελσαλβαδόρ ως πρώτο θέμα και το δεύτερο θέμα θα είναι το προσφυγικό που είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Όσον αφορά τώρα τα ταξίδια, ε, εκκρεμούν βεβαίω, ε, δεν είναι με ευθύνη του Προεδρείου. Είναι γεγονό ότι ακυρώθηκαν γιατί συνάδελφοι οι οποίοι είχαν δηλώσει για του δικού του λόγου και για τι ε, αυξημένε υποχρεώσει που είχαν ε, δεν καταφέραν να έρθουν σε αυτό το ταξίδι, άρα το ακυρώσαμε. θα συζητήσουμε. Θέλω να σα ενημερώσω βεβαίω για να είμαι και δίκαιη, γιατί με την Κούβα <laughs> δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό που που γνωρίζω είναι ότι έχουμε μια ανοιχτή συνεννόηση με την κυρία Κοϊκοτσέα όσον αφορά τη συζήτηση για το πώς θα οργανώσουμε αυτό το ταξίδι, αν αποφασίσουμε τελικά ως ε, αντιπροσωπεία να πάμε. Και νομίζω ότι εδώ είμαστε για να το κουβεντιάσουμε, αν θέλετε, και στην επόμενη συνεδρίαση, όποτε εσείς νομίζετε. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν τις κυρίες και τους κυρίους. Να σας θυμίσω ότι είναι στις 28 Ιουνίου η επόμενη συνεδρίαση εδώ. Να σας ευχαριστήσω όλους για την υπομονή σας σήμερα, να ευχαριστήσω και τους μεταφραστές μας και να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.